Ähm, Κυρίες και κύριοι, θα εκπροσωπήσω μόνο εγώ την ομάδα μου. Αναμένουμε άλλο ένα μέλος της ομάδας. Δεν θέλουμε όμως να χάσουμε χρόνο, οπότε σας καλωσορίζω στην ενημέρωσή μας. Είμαι η Γκάβιτ Τσίμερ, πρόεδρος της ομάδας. Δίπλα μου είναι ο κύριος Μιγκέλ Βιέγκας, ο οποίος ε, μετά από μένα θα μιλήσει για την συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Κάνω μια εισαγωγή. Ξέρετε ότι έχουμε το απόγευμα τη συζήτηση για την Τουρκία που είναι στο επίκεντρο. Είναι μια συζήτηση η οποία ξεκίνησε και από την ομάδα μας άμεσα μάλιστα μόλις ακούσαμε για το νέο κύμα συλλήψεων ε, που αφορούσε και την ηγεσία του ΧΑΝΤΕΠΕ αλλά και ε, ακόμη περισσότερους δημοσιογράφους ε, και μέλη της αντιπολίτευσης και θεωρήσαμε ότι έπρεπε να κινηθούμε άμεσα ως κοινοβούλιο. Ε, φαίνεται ότι οι πρώτες προσπάθειες ε, συνεννόησης με την ηγεσία του Κοινοβουλίου και άλλες ομάδες ε, δεν μπόρεσαν να οδηγήσουν σε γρήγορη αντίδραση για να στείλουμε μια αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στην Τουρκία. Εμάς η πρόθεσή μας ήταν να λάβουμε μια γρήγορη υπόσχεση από τις τουρκικές αρχές ότι οι βουλευτές από όλες τις ομάδες θα μπορέσουν να ταξιδεύσουν και να έρθουν σε επαφή με τους συλληφθέντες. Έγιναν προσπάθειες τις τελευταίες μέρες να, πήγαν να πάνε κάποιοι βουλευτές μεμονωμένοι όμως. Δεν υπήρχε δυνατότητα όμως να έχουν επαφή με τους συλληφθέντες. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ πως είναι σωστό να θέσουμε την δεύτερη επιλογή, δηλαδή να γίνει μια συζήτηση στο Κοινοβούλιο ακριβώς για να δούμε την σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Αυτό μας ενδιαφέρει εμείς. Έχουμε πει πολλές φορές ποια είναι η δική μας η κριτική απέναντι στην τωρινή τουρκική κυβέρνηση, ότι θεωρούμε ότι από... με βάση το πώς ε, κύλησαν τα πράγματα μετά το πραξικόπημα. Είχαμε μία αντιστροφή της κατάστασης και το εκμεταλλεύτηκε για να κάνει το δικό του αντιπραξικόπημα. Ο Τούρκος Πρόεδρος με χιλιάδες συλλήψεις και λέμε ότι αυτή η πτυχή πρέπει οπωσδήποτε να καταργήσει την συμφωνία με την Τουρκία και να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια δική της μεταναστευτική πολιτική. Δεν μπορεί να διαπραγματεύεται με ένα τέτοιο καθεστώς μια συμφωνία και μετά να λέει πρέπει να συμφωνήσει και να εξαρτάται και να είναι τόσο ανοιχτή στην κριτική. Να μην ε, μπορεί δηλαδή να αρθρώσει δική της ε, δικό της κριτικό λόγο. Βλέπω με τι διατυπώσεις ε, προσπαθούν ε, στο Βερολίνο και αλλού να πούν ε, ότι δεν είναι πράγματα αυτά. Είναι σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει συνεργασία με ένα καθεστώς το οποίο περιφρονεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους βασικούς κανόνες της ε, δημοκρατίας. Επίσης, εμείς είμαστε υπέρ του να παγώσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Δεν λέμε να διακοπούν, να παγώσουν μέχρι να υπάρξουν, να αλλάξουν οι συνθήκες. Θέμε έτσι λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι το θέμα επί της αρχής δεν είναι ότι έχουμε πρόβλημα η Τουρκία να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ και χρόνια προσπαθούσαμε εμείς να ξεκινήσουν και να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Αλλά βεβαίως ε, αυτό το οποίο δεν μπορούμε να αποδεχτούμε είναι το να παριστάνουμε ότι τα βήματα προς τα πίσω που έχουν γίνει στην ε, Τουρκία να κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε και να καθορίζουμε ξανά τους κανόνες για ένταξη. Ζητάμε λοιπόν την αποκατάσταση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, την απελευθέρωση συλληφθέντων, πολιτικών και δημοσιογράφων ως βασική προϋπόθεση για την συνέχεια των διαπραγματεύσεων και υπενθυμίζουμε κιόλας ε, και θα συζητηθεί και σήμερα ε, τις κυρώσεις κατά των τουρκικών αρχών. Δεν θέλουμε κυρώσεις ε, που θα πλήξουν τον τουρκικό λαό, αλλά θέμε να ξεκαθαρίσουμε πως αυτοί οι οποίοι μαζικά και συνεχώς και με αλαζονία περιφρονούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου ε, θα πρέπει να, να πούμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να τα παρακολουθεί απλώς αυτά. Πρέπει να πει πως ε, αυτά δεν ταιριάζουν με τη δική μας ηθική και τις δικές μας ε, αξίες. Και ακριβώς θα πρέπει να δούμε και τα άλλα γεγονότα. Η Τουρκία ζήτησε συγγνώμη για την κατάρριψη ενός, τουρκικού, ενός ρωσικού αεροσκάφους και... Ακούμε τώρα για τον νόμο ότι οι βιαστές θα απαλλάσσονται αν παντρευτούν το θύμα τους να υπάρξει τουλάχιστον μια αντίδραση σε αυτά τα πράγματα. Όλα αυτά για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία απαιτούμε και λέμε πως είναι σημαντικό να υπάρξει αυτή η πίεση. Ελπίζω λοιπόν η συζήτηση αυτή να αυξήσει την πίεση στην Τουρκία. Να ξεκαθαρίσουμε ότι οι αιματηρές συγκρούσεις ε, στις κουρδικές περιοχές επίσης είναι απαράδεκτες ε, και ζητάμε επίσης ε, η κυβέρνηση του ΑΚΠ να μην επαναφέρει την θανατική ποινή και να τηρήσει τα όσα έχει αναλάβει ως δεσμεύσει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παρ' όλα αυτά, το Κοινοβούλιο δεν πρέπει να διακόψει τις συνομιλίες με το τουρκικό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα συναντώνται με Τούρκους συναδέλφους τους ε, για να μπορέσουμε έτσι να ασκήσουμε κάποια επιρροή και να πούμε ποιες είναι οι δικές μας οι απαιτήσεις και τελικά να παραμείνουμε σε αυτόν τον διάλογο με την ε, Τουρκία. Αυτά από εμένα. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον Μιγγέλ Βιέγκας. Bom dia. Nós tivemos esta semana a Καλημέρα. Εμεί αυτή την εβδομάδα κάναμε τη συζήτηση επικεντρωμένη σε δύο πτυχέ πολύ σημαντικέ. στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και το δεύτερο μια νέα οδηγία διοικητική συνεργασία με σκοπό την εισαγωγή ζητημάτων που σχετίζονται με την νομιμοποίηση εσόδων από παρανομές δραστηριότητες. Όσον αφορά το ευρωπαϊκό εξάμεινο, τώρα ξεκινά επίσημα ένας νέος κύκλος οικονομικής διακυβέρνησης, ε, η πολιετής προοπτική της ανάπτυξης, ε, ε, και ο σχετικό μηχανισμό αποτελούν ένα πρώτο βήμα οικονομικού κύκλου που θα οδηγήσει στην έγκριση του προπολογισμού του 2018. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για να τεθούν τα πρώτα θεμέλια πάνω στα οποία σύμφωνα με τους κανόνες οι εθνικές κυβερνήσεις υποτίθεται ότι θα βασιστούν για να ξεκινήσουν το δικό τους προπολογισμό. Όσον αφορά την έκθεση δεν βλέπουμε κάτι νέο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμένει στη στρατηγική που βασίζεται στις διαρθρωτικές επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις και στη δημοσιονομική πειθαρχία, δηλαδή δεν καταλαβαίνει το πόσο δεν συμβαδίζουν αυτές οι τρεις προτεραιότητες ε, πρακτικά. Ε, συνεπώς ε, δεν είναι δυνατόν να ξεκινάμε πολιτικές οικονομικές ανάπτυξης σε ένα πλαίσιο λιτότητας που έχει επιβληθεί στο πλαίσιο της δημοσιονομικής πειθαρχία. Έξω και τα λοιπή αποτελέσματα στο μέτωπο της οικονομίας. Ελαφριά βελτίωση σημείωσε η ανάπτυξη, αλλά πραγματικά πολύ μικρή παραμένουν τα σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα της ευρωπαϊκής οικονομίας με υψηλούς δείκτες φτώχειας, ποσοστά ανεργίας και ειδικότερα όσον αφορά τι νεότερες μερίδες του πληθυσμού. Από την άλλη έχουμε και κάτι νέο σε σχέση με την πολύ ιδιαίτερη κατάσταση της πορτογαλικής οικονομίας. Όπως θα ξέρατε, τον Οκτώβριο του 2015 είχαμε εκλογές οι οποίες οδήγησαν ε, στην εφαρμογή μιας σειρά πολιτικών οι οποίες ε, ανέτρεψαν πολλά από τα μέτρα τα οποία είχαν επιβληθεί από την Τρόικα ε, αύξηση της, του ελάχιστου μισθού, μείωση των ωραρίων εργασίας, μείωση του φορολογικού βάρους για την εργασία. Δόθηκε τέλος σε ορισμένες ιδιωτικοποιήσεις και αυτό οδήγησε σε μια εκδίκηση, σε μια ε, απειλή εκ μέρους της Κομισιόν που θεωρούσε πάντα ότι αυτά αποτελούσαν κινδύνους για τη σταθεροποίηση των, και την εξηγένση των δημοσίων οικονομικών. Εμείς είδαμε λοιπόν ότι αντίθετα από τα πόσα ισχυριζόταν η Κομισιόν, η πορτογαλική οικονομία αυτή τη στιγμή σημειώνει αύξηση πολύ μεγαλύτερη από ό,τι παλιότερα. Και για πρώτη φορά στην ιστορία το έλλειμμα θα είναι κάτω του 3%, δηλαδή ακριβώς το αντίθετο από αυτό που είχε προβλέψει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό λοιπόν αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο ε, κατά μία έννοια αποδεικνύει ότι η πολιτική λιτότητας ε, δεν είναι τόσο σωστή και δείχνει ότι είναι δυνατόν να μην ακολουθήσει κανείς αυτά τα μέτρα, να τα αντιστρέψει και να οδηγήσει μια άλλη οδό ώστε να επανεκκινήσει όχι μόνο την οικονομία αλλά και για μεγαλύτερα έσοδα. χωρίς αυτό να σημαίνει ανεύθυνη πολιτική όσον αφορά τα δημόσια, ε, τις δημόσιες δαπάνες. Αυτό όμως ε, δεν αναγνωρίστηκε. Βλέπουμε να συνεχίζεται ένας οικονομικός έλεγχος ως μέσο επιβολής μιας πολιτικής και μιας σειράς προτεραιοτήτων νεοφιλελεύθερων σε οικονομικά θέματα εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, από αυτή την άψη λοιπόν Τα όσα παρατηρούμε στην πορτογαλική οικονομία είναι πολύ ενδιαφέροντα και πολύ ε, σημαντικά. Ωστόσο, δεν αλλάζουν τη θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εξακολουθεί να πιστεύει ότι ε, ο οικονομικό έλεγχο είναι ένα μέσο ελέγχου τη οικονομία και των πληθυσμών, αλλά πάνω απ' όλα ένα εργαλείο επιβολή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ουσιαστικά να αφαιρέσει αρμοδιότητες από το κράτος, οι κοινωνικές, οι οικονομικές επίσης. Σήμερα το πρωί πέραν αυτού συζητήθηκε και μια τροποποίηση της οδηγίας του 2011 με στόχο την παρεμβολή στη διοικητική συνεργασία ε, για το Δημοσιονομικό Σύμφωνο των Κρατών Μελών. Αυτό σχετίζεται με την ε, καταπολέμηση της νομιμοποίησης όταν παράνομες δραστηριότητες. Για αυτή την τροποποίηση εμείς έχουμε θετική άποψη για αυτή την τροπολογία και θεωρούμε ότι παρόλα αυτά οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να ανταλλάσσονται αυτόματα ώστε αυτή η τροπολογία να ε, οδηγήσει σε μια σοβαρή ε, επί της ουσίας αλλαγή. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τις χώρες ελεύθερες να αποφασίζουν κατά πόσο θέλουν να πραγματοποιήσουν ανταλλαγή δεδομένων ή όχι. Τα δεδομένα αυτά, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να ανταλλάσσονται αυτόματα. Και με μια περαιτέρω λοιπόν τροπολογία επί της τροπολογίας που υποβλήθηκε για την έκθεση, εμείς ευθυγραμμιζόμαστε με τα όσα θεωρήθηκαν απαραίτητο. <clears throat> Ωραία. Λοιπόν, άρα θα ακούσουμε και την κυρία Κωνσταντίνα Κουνβά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και από μένα. Σήμερα θα σας μιλήσω για ένα θέμα το οποίο είμαι σκιώδης συγκήτρια την πολιτική ομάδα της Γκουέντζελ στην Επιτροπή Γυναικών ΦΑΜ. Πρόκειται την ενδιάμεσα έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Τι είναι η σύμβαση αυτή. Ουσιαστικά, το πρώτο στο είδο του, δεσμευτικό, διεθνή νομικό εργαλείο για να εξαλείψει και να προλάβει τη βία κατά των γυναικών επικεντρώνεται δηλαδή σε τέσσερα βασικά θέματα. Την πρόληψη της βίας, την προστασία των τιμάτων, την δίωση των δράστων και την παρακολούθηση. Όμως είναι σημαντική και ένα άλλο λόγο, γιατί προβλέπει την ανάπτυξη ενός συστήματος παροχής ασύλου με βάση το φύλλο πάνω στη βάση του ότι η υποχρέωση προστασίας περιλαμβάνει το δικαίωμα διεθνούς προστασίας. Γυναίκες θύματα βίας μπορούν να ζητήσουν προστασία σε άλλο κράτος όταν το δικό τους αποτυχάνει να τους την προσφέρει. Όταν μιλάμε για έμφυλη βία, μιλάμε για το πιο δεδομένο έγκλημα στον κόσμο, που πλήττει τη ζωή, την αξιοπρέπεια και την ελευθερία του μισού πληθυσμού της γης. περνά όλους τους πληθυσμούς της χώρας και της κοινωνίας μας. Υπάρχει και εξακολουθεί να υπάρχει η βία λόγω φύλου. Και δεν συμβαίνει κάπου μακριά μας. Ένα στις τρεις γυναίκες στην Ευρώπη γίνεται θύματα βίας, σεξουαλικής, φραστικής, σωματικής ή ψυχολογικής και ασκείται όχι πάντα πίσω από κλειστές πόρτες των οικοκυριών. Σκεφτείτε πως σχεδόν οι μισές γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δηλώσει πως έχουν υποστεί κάποια μορφή βίας στο χώρο που εργάζονται. Δυστυχώς, ο φόβος έγινε κανόνας και σε συνδεσμό με τη γενικότερη οικονομική κρίση επιβλήθηκε η σιωπή στη βάση χιλιάδων χιδαίων εκβιασμών με τυχόν και χάσουν την δουλειά τους ή δεν ανέβουν ιεραρχικά. Τι κάνουμε όμως εμείς εδώ, εκτός από το να σας ενημερώνουμε με στατιστικά δεδομένα και επαναλαμβάνοντας πράγματα γνωστά εδώ και χρόνια. Αφενός πιέζομαι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία με προφορική ερώτηση που συντάξαμε καλούμε να αναπτύξει αύριο στην Ολομέλεια για το τι πρόκειται να κάνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολη. Περιμένουμε να ακούσουμε τι μέτρα η πρωτοβουλία θα λάβει για να γίνει πιο γρήγορα η επικύρωση της Σύμβασης τόσο από την ίδια όσο από άλλα κράτη-μέλη της Ευρώπης αλλά και πιο συγκεκριμένα μέτρα έχει σκοπό να λάβει για να ενισχύσει τα κράτη-μέλη στις προσπάθειες τους να εξαλείψουν τη βία ανάντια στις γυναίκες. Από την άλλη, προετοιμαζόμαστε να συντάξουμε την ενδιάμεση έκθεση για την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, έναν φάκελο που τρέχουν στην Επιτροπή ΦΑΜ και εγώ από την πλευρά της ΓΟΕ και η Επιτροπή για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα με την Μάλιν Μπιόρκ από την ΚΟΕ. Σηκώνουμε μανίκια και προσπαθούμε να δούμε τι άλλα επιχειρήματα τα φέρουμε για να καταφέρουμε να πάρτουν μέτρα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο στα κράτη-μέλη. Γιατί τα λογικά επιχειρήματα, ξέρετε, δεν, δεν τα ακούν. Μερικές φορές, όσες και όσους μιλάμε για έμφυλες βία, μας αντιμετωπίζουν με κινησμό, σαν να είμαστε γραφικοί και αυτό μας, μας προβάλλουν σαν επιχείρημα για την λήψη μέτρων Συγγνώμη. Και αυτό που μας προβάλλουν σαν επιχείρημα για τη λήψη μέτρων για τα λεφτά. Το υψηλό κόστος εφαρμογής όπως χαρακτηριστικά λένε. Ένα λοιπόν από τα πράγματα που τα βάλουμε μέσα στην έκθεση είναι πως τα κράτη-μέλη δεν συνυπολογίζουν εκτός από τα ψυχολογικό κόστος για τους πολίτες το κόστος που προκύπτει από την άσκηση βίας τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνία γενικότερα. Οι άμεση και έμεση δαπάνε που προκύπτουν όταν ασκείται βία ανέρχονται σήμερα στα 47 μέλη του Συμβούλου της Ευρώπης στα 34 δισεκατομμύρια ευρώ και ελπίζουμε με αυτό το επιχείρημα να πείσουμε τις κυβερνήσεις που συνήθως είναι πιο ευαίσθητες στον ήχο του χρήματος να προχωρήσουν πιο γρήγορα στην κύρωση. Σε ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαστε διάθεση σε ετυχόν ερωτήσεις που έχετε να κάνετε σε εμάς. Uh, Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνα Καμπρίλ και Μιγγέλ. Τώρα ε, δίνουμε το λόγο ε, στους περιστάμενους για ερωτήσεις. Ε, έχουμε περιορισμένο χρόνο, παρακαλώ να είστε σύντομοι. Euh, Καλημέρα κυρία Πρόεδρε. Όπως φαίνεται όλες οι πολιτικές ομάδες συμφωνούν ε, στο πράγμα των σχέσεων με την Τουρκία πώς ε, θα επηρεαστούν οι οικονομικές και εμπορικές μας σχέσεις ε, και οι σχέσεις με την Τελωνιακή Ένωση και τα διαρθρωτικά ταμεία. Όπως φαίνεται, για αυτή την πτυχή οι απόψεις μεταξύ των ομάδων δίστανται. Ποια είναι η δική σας άποψη, τι αναμένετε πιο συγκεκριμένα από το Συμβούλιο και από την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Υποθέτω πως δεν μιλάτε για την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, μιλάτε για την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και τη γενικότερη σχέση. Κοιτάξτε, θεωρώ πως ε, έχουμε διαφορές ε, στα συγκεκριμένα πράγματα που ζητάμε. Παραδείγματο χάρη, να σκεφτούμε ότι δεν, είναι, ε, δεν ζητάνε όλες οι ομάδες να σταματήσει η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Δεν τον ζητάνε όλες. Και δεν λένε ότι δεν μπορεί να βασίζεται η μεταναστευτική μας πολιτική σε ένα καθεστώς το οποίο παράγει περισσότερους πρόσφυγες από τις κουρδικές περιοχές, που τους διώχνει από τα σπίτια, από τα χωριά τους, ε, τις περιοχές τους κτλ. Δεν είναι δυνατόν και δεν μπορεί να περιμένουμε η Τουρκία με την αντίληψη που έχει για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, να καθορίζει μια τέτοια πολιτική. Εμείς λοιπόν θα παραμείνουμε σε αυτό το αίτημα. Θέλουμε να μας πει ξεκάθαρα η Κομισιόν τι γίνεται με τα λεφτά τα οποία υποτίθεται ότι ήταν για την ενταξιακή διαδικασία και τώρα ε, πηγαίνουν ε, για τη φροντίδα των προσφύγων εντός της ε, Τουρκίας, στο πλαίσιο ακριβώς αυτής της συμφωνίας. Εδώ πέρα θέλουμε η Κομισιόν... Βλέπουμε ότι η Κομισιόν πρέπει να τα πει ξεκάθαρα. Υπάρχει ακόμα κάποια πιθανότητα ένταξης ή αλλιώς γιατί διοχέτευσε αλλού τα λεφτά. Και για να το ε, αντιστρέψω πρέπει και για όλους και για την Τουρκία να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Πού πηγαίνουμε επιπλέον λέμε ότι ε, κυρώσεις βεβαίως θα αφορούν προσωπικά πολιτικούς άτομα και μέλη της ε, τουρκικής ε, κυβέρνησης. Αν σκεφτούμε, παραδείγματο χάρη, πόσο γρήγορα επέβαλε κυρώσεις κατά της Ρωσίας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και είχαμε μετά παράλογες ε, λίστες κυρώσεων και από τις δύο πλευρές. Γιατί μετά κλιμακώθηκε η κατάσταση. Ή έχουμε λίστες κυρώσεων από εθνικά κοινοβούλια ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εμείς από την άλλη πλευρά είχαμε άτομα στη λίστα τα οποία αναρωτιέμαι ξαφνικά αυτοί είναι υπεύθυνοι για την προσάρτηση της Κρυμαίας. Τι σχέση έχουν. Δηλαδή έχουν γίνει τόσα πολλά πράγματα λανθασμένα σε σχέση με τη Ρωσία, ώστε εδώ πέρα σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ακριβώ να στοχεύσουμε άτομα τα οποία είναι άμεσα υπεύθυνα για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διώξει και βασανιστήρια στην Τουρκία. Να υπάρξει δηλαδή μια λίστα κυρώσεων ε, με πολιτικά πρόσωπα ε, που χρησιμοποιούν τέτοιε μεθόδου. Τότε έχει νόημα. Δεν είμαι τώρα διατεθειμένη και δεν είμαι υπέρ αυτή τη στιγμή να περιοριστούν οι οικονομικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ούτε και για, την, ούτε και για τη Ρωσία όμως ήμουν. Ε, έχω επί της αρχής επιφυλάξεις κατά τέτοιων κυρώσεων. Ευχαριστώ Καμπή. Μια τελευταία ερώτηση. Χθε ήταν εδώ η μητέρα του δολοφονημένου από την Χρυσή Αυγή ε, Μάγδα Φίσα για να ενημερώσει την ΚΟΕ ε, για την πορεία της δίκης και τα προβλήματα μέσα και έξω από την αίθουσα. Ε, η πρώτη μου ερώτηση λοιπόν είναι ποια είναι η αίσθησή σας και τι προτίθεται να κάνει η ΚΟΕ για ε, την κατάσταση αυτή που επικρατεί στην Αθήνα. Και το δεύτερο είναι, με αυτή την αφορμή, μήπως έχετε κάποιο νέο σε σχέση με τη χρηματοδότηση της Χρυσής Αυγή και άλλων ε, φασιστικών και ρατσιστικών κομμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπήρξε μια προσπάθεια να, εξεταστεί αυτό το ζήτημα. Έχουμε κάποιο νέο σχετικά με αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, τώρα θα από την δεύτερη ερώτηση ότι ακόμα εξετάζουμε, έχουμε ενημερωθεί, το ψάχνουμε ακριβώς πώς γίνεται. Ε, πιστεύω ότι αν είναι κάτι παρόνιμο θα το, το βρούμε. Ε, και όπως και να είναι θα, θα, το, το δημοσιεύσουμε. Για να ξέρει ο κόσμος πώς γίνεται η χρηματοδότηση. το άλλο ότι είναι, ήταν μια πρώτη, ένα πρώτο βήμα αυτό σαν δράση της ΓΟΕ για να αντιμετωπίζουμε την δίκη αυτή και να τους βοηθήσουμε. Τώρα κάνουμε προγραμματισμό, βάζουμε ιδέες, ε, πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε και από επιτροπές μέσα στην Ευρωβουλή και εμείς ε, σαν ε, ομάδες από διάφορες χώρες της Ευρώπης να το στηρίξουμε και να προβληθεί το πρόβλημα με τη Χρυσή Αυγή σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνκα. Αυτά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώ. Ευχαριστώ σε όλου για, για τον χρόνο σα και τι τελευταίε αλλαγέ του προγράμματο, τι αλλαγέ τη τελευταία στιγμή. Ε, αν έχετε οτιδήποτε άλλο, παρακαλώ απευθυνθείτε απευθεία στου βουλευτέ.